Αξιότιμοι πρόεδροι των Επιτροπών, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, είναι προνόμιο για μένα να επανέρχομαι εδώ για δεύτερη φορά ως υποψήφια επίτροπος. Θυμάμαι σαν χτες την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ για την ακρόασή μου, μετά από την οποία προχώρησα σε ιδιαίτερα καρποφόρα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βασιστήκαμε σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Εφόσον επιβεβαιωθώ στο χαρτοφυλάκιό μου, προσβλέπω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μέσα στο ίδιο πνεύμα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά, αλλά και ειδικότερα με τις τρεις επιτροπές που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Αυτή τη φορά βρίσκομαι εδώ ως υποψήφια αντιπρόεδρος για τον προπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους. Καταλαβαίνοντας πάρα πολύ καλά πόσο ζωτική σημασία είναι να κινητοποιήσουμε τους οικονομικούς μας πόρους και τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα τις υποσχέσεις που δώσαμε στους Ευρωπαίους. Και νομίζω ότι κεντρικό σημείο στη δουλειά μου, εφόσον επιβεβαιωθώ, είναι να καθορίσω προτεραιότητες βάσει των δυνατοτήτων των οικονομικών που έχουμε και να αποδώσουν οι πόροι αυτοί όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια νοοτροπία επιδόσεων και να λογοδοτούμε στους πολίτες οι οποίοι πληρώνουν τελικά για τη δουλειά που κάνουμε εμείς και οι οποίοι πρέπει να υποφελούνται από τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς αλλά και οι συναδελφοί μου, όπως το ακούσαμε και από τους πρέδρους πριν από λίγο, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να απαντήσουμε στα εξή ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι πετυχαίνουμε με κάθε ευρώ που δαπανά η Ευρώπη προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολίτες μας και τις οικονομίες μας. Μπορούμε να αποφύγουμε με τους έλεγχους μας χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων να καταλήξουν σε κατάχρηση. Μπορούμε να το λέξουμε αυτά καλά και να αποφύγουμε την κατάχρηση. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το προσωπικό μας, ώστε να φτάσει την αριστεία να έχει υψηλά το ηθικό γιατί του δίνει ικανοποίηση η δουλειά που κάνει. Στα πλαίσια λοιπόν των τόσο δύσκολων καιρών που ζουν τόσοι πολίτες μας, εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο γίνεται πιο σοφά και να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της κρίσης που κρατάει τόσο καιρό, αποτελέσματα που έχουν πλήξει τον ανταγωνισμό, τις ε, αγορές απασχόλησης και την ίδια την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμό μπορεί να το πετύχει αυτό, μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας, μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη και να τη δει σε μια δύναμη του καλού. Ξεκινάμε από μια καλή βάση και αυτό είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 ένα 3 ευρώ περίπου επενδύσεις για τα επόμενα 7 χρόνια για βελτίωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και βελτίωση της καθημερινής μας ζωής. Δεν πρόκειται για αφηρημένα νούμερα. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει άμεσες επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων. Σημαίνει δουλειά για περίπου 600.000 ανθρώπους σε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχής και σημαίνει και δουλειά για εκατοντάδε. χιλιάδες άλλους επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν υποδομές και υλικά. Σημαίνει και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για 4 εκατομμύρια ε, φοιτητέ, οι οποίοι θα αποφεληθούν από το Erasmus ε, Συν, το πρόγραμμα αυτό Erasmus. Και αυτό σημαίνει ότι ο τομέας για τον οποίο θα είμαι εγώ αρμόδια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και μπορεί να κάνει διαφορά και ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο για πολλά θύματα σε χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση σήμερα ή που υποφέρουν από φυσικές καταστροφές. Αλλά αυτό για να υλοποιηθεί χρειάζεται πολλή δουλειά και μερικές καλές ιδέες έχουν ε, ακουστεί και τις έχετε συζητήσει κι εσείς όταν ψηφίσατε το σχέδιο προπολογισμού για το 2015. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεφορτωθούμε τις οφειλές που έχουμε, να τις πληρώσουμε. Έχετε δει εξάλλου ότι και η σημερινή Επιτροπή φάνηκε με την επιστολή του Πρόεδρου Μπαρόσο στους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων και στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, φαίνεται λοιπόν ότι τους απασχολεί ήδη αυτό το πρόβλημα πολύ. Και βρίσκεται πάνω-πάνω στις υποχρεώσεις που μου έχει αναθέσει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ, εφόσον επιβεβαιωθώ. Από την πρώτη μέρα λοιπόν που θα αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα θα φροντίσω να συνεργαστώ με τον Επίτροπο Ντόμινικ για να πετύχω στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για το σχέδιο προπολογισμού 2015 αλλά και για τους διορθωτικούς προπολογισμούς 2014 ώστε πια αυτή η χιονοστιβάδα απλήρωτων λογαριασμών να μειωθεί. Και είμαι πεπισμένη ότι αν δεν το κάνουμε αυτό τότε σκάβουμε το λάκκο μας. Διότι σημαίνει ότι αναβάλλονται προβλήματα τα οποία αν λυνόντουσαν θα δημιουργούσαν θέσεις απασχόλησης και θα καταλήξει ο λογαριασμός να είναι ακόμα πιο ακριβώς για μας γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε ε, πρόστιμα και υψηλού τόκου υπερημερία. Κάτι το οποίο εξάλλου θίγει και την ίδια μα τη φήμη και την εξοπιστία. Είναι όμω ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί. Και μπορεί να λυθεί απλώ και μόνο εφαρμόζοντα την ευελιξία. Ευελιξία που εσεί ίδιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θελήσατε και πετύχατε μετά από σκληρό αγώνα. Όλοι τελικά συμφώνησαν. Δεν ζητάμε περισσότερα χρήματα για πληρωμές, από ό,τι έχουμε στο τωρινό πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που ζητάμε είναι περισσότερα χρήματα σήμερα, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις. όπως για παράδειγμα το που υπάρχουν περισσότερα πλήρω λογαριασμοί για την συνοχή, επειδή επιταχύθηκαν κάποια προγράμματα, δόθηκαν προκαταβολές και υπάρχει βέβαια και ε, το θέμα της Ουκρανίας. Αλλά πέρα από αυτές τις άμεσες προτεραιότητες υπάρχουν και άλλα θέματα για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα η μεταρρύθμιση των, ε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που η αναθεώρηση αυτή στα μέσα του δρόμου θα γίνει το 2016 και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες προκειμένου ο ευρωπαϊκός ε, προϋπολογισμός να προσανατολιστεί περισσότερο στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και θα μας επιτρέψει αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις που θα έχουν εμφανιστεί. Πώς όλα αυτά τώρα θα ευθυγραμμιστούν με τον οικονομικό κύκλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι σημαίνουν αυτά προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τις ειδικέ ανάγκες της Ευρωζώνης. Μόλις αναλάβει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η σημερινή απερχόμενη επιτροπή, της οποίας είμαι εγώ μέλος, θα κάνει προτάσεις για την αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και στην ομάδα υψηλού επίπεδου υπό την Προεδρία του καθηγητή Μάριο Μόντι να προβληματιστούμε και να λάβουμε υπόψη μας και τις προπτικές που υπάρχουν για να αναθεωρηθεί το σύστημα ιδίων πόρων μας και να προσπαθήσουμε να βρούμε νέους δρόμους για το μέλλον. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να συζητηθεί και στην προσωρινή μεταρρύθμιση αλλά και κυρίως στην προετοιμασία των νέων, του νέου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου συζητήσεις που θα ξεκινήσουν τον ε, Ιανουάριο του 2018. Μεταξύ άλλων προτάσεων θα φροντίσω να λάβω υπόψη μου και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συνεργαστώ μαζί του όπως επίσης και με τους άλλους εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσει αυτές και να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά μας καλύτερα και ότι αλλάζουμε νοτροπία δαπανών προκειμένου να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα. Πρέπει να αποδείξουμε δηλαδή ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν έχει απλώς καλύτερη απόδοση, αλλά μεγάλη απόδοση για όλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν οι επιδόσεις μας όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων και σημαίνει επίσης και περισσότερη μόχλευση από ό,τι είχαμε κατά το παρελθόν. Κάνοντας αλλαγές ε, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε καινοτομίε στα οικονομικά μέσα που διαθέτουμε. Παράδειγμα, το ομόλογα έργου που πολλαπλασιάζουν το αποτέλεσμα των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 40 τέτοιου είδους καινοτόμα οικονομικά μέσα θα έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του νέου πακέτου επενδύσεων των 300 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις πολιτικές του κατευθυντήριες γραμμές. Επενδύοντας λοιπόν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε προγράμματα τέτοια θα είναι μεγάλο κέρδος. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, για παράδειγμα, θα αυξήσει τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην ενέργεια, το οποίο με τη σειρά του θα δώσει νέα όθηση σε επενδύσεις, σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θα, μειωθεί, θα μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα καταπολεμηθεί καλύτερα η κλιματική αλλαγή και θα μας βοηθήσει επίσης να μειώσουμε και την ενεργειακή μας εξάρτηση. Πολύ σημαντικό μέρος των δράσεών μας για τον καλύτερο τρόπο δαπανών είναι η αντιμετώπιση των ε, καταχρήσεων των πόρων. Μια πολύ σημαντική στιγμή στη διαδικασία αυτή είναι η απαλλαγή, όπου αξιολογούμε κατά πόσο τα κονδύλια μας έχουν δαπανηθεί σωστά. Και έχουμε προγράμματα τα οποία μας βοηθούν να δαπανούμε σωστότερα, με λιγότερα σφάλματα και με πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Όμως παρόλα αυτά μένει πολλής δρόμος ακόμα και χρειάζονται επιπλέον βελτιώσεις για τη συμμόρφωση, κάτι το οποίο είναι βασικός μας στόχος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη λογοδοσία των χωρών μελών και των διεθνών μας εταίρων. Μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα επίσης για να απλοποιηθούν οι κανόνες αναφοράς, όπως ε, επίσης και αξιολόγησης κινδύνου. Είναι πράγματα όμως που πρέπει να γίνονται καλύτερα κατανοητά, γιατί τότε θα μπορούν όλοι να συμμορφωθούν και καλύτερα. Άρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα όπου θα επικεντρώνουμε την προσοχή μας εκεί που υπάρχουν οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι. Θα συνεργαστώ λοιπόν στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις χώρες μέλη, με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, με τις Εθνικές Ελεκτικές Αρχές και με τους διεθνείς μας εταίρους. Θα στηρίξω μία Όλαφ ανεξάρτητη και ισχυρή προκειμένου να προστατεύει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απάτες και οι καταχρήσεις κλέβουν ουσιαστικά χρήματα από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και καταστρέφουν το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κάτι το οποίο δεν θα ανοιχτώ. Και για το σκοπό αυτό θα ήθελα πολύ να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι κλιματικές ενέργειες και οι καταχρήσεις δημοσίου χρήματος. Τέλο, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο προσωπικό μα, γιατί τίποτα από αυτά τα οποία σα ανέφερα μέχρι τώρα δεν θα γίνει πραγματικότητα αν δεν έχουμε αριστεία στο προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των άλλων θεσμικών οργάνων. Ζούμε σε εποχές μεγάλου ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν επί συνεχούς βάσεως να βελτιωνόμαστε αν θέλουμε να έχουμε πρώτης τάξεως υπαλλήλου. Και αυτό είναι κάτι που ως μήνυμα θα το πω και θα το ξαναπώ. Και έχει πολύ σημασία να ληφθεί υπόψη στη δίκηση γενικότερα. Πρώτα απ' όλα πρέπει η ευρωπαϊκή απασχόληση να είναι, απασχόληση δηλαδή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να είναι κάτι ελκυστικό. Και να βοηθούμε επίσης το προσωπικό να καλυτερεύει. Να διασφαλίσουμε και τη συμμετοχή των γυναικών εξίσου όπως και των ανδρών. Έτσι θα έχουμε έμπειρο προσωπικό τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω στη δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού και στην ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Και θα φροντίσω να πετύχω το 40% που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος γυναίκες σε υψηλά και σε μεσαία αξιώματα διοικητικά. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε την ευελιξία και την κινητικότητα στο προσωπικό μας και να χρησιμοποιήσουμε τη δομή της νέας επιτροπής που επιτρέπει το προσωπικό να αλλάζει θέσεις πιο εύκολα. Τρίτον, πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο αποδοτικοί στη χρήση του προσωπικού. Δεν πρέπει να αφήσουμε καμία πέτρα χωρίς να τη σηκώσουμε να δούμε τι υπάρχει από κάτω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι μια δυνατή και αποτελεσματική ομάδα. Χρήματα και άνθρωποι έχουν τεράστια σημασία προκειμένου η ζωή των Ευρωπαίων να γίνει καλύτερη. Αυτό όμως που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι οι αξίες. Οι αξίες εκείνες οι οποίοι μας έχουν κάνει αυτούς που είμαστε, που μας βοηθούν να ξεπερνάμε τις διαφορές και να μην μείνει κανείς ξεχασμένος. Έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μπορούμε να νοιαστούμε για τους πιο ευάλωτους τόσο στις χώρες μας όσο και αλλού. Και ακριβώς εξαιτία των ε, αξιών αυτών είμαι περήφανη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τιμή για μένα που ζητάω την εμπιστοσύνη σας για να αναλάβω το χαρτοφυλάκιό μου. Ευχαριστώ πολύ.